Dámy Κυρίες και κύριοι, κηρύττω την επανάληψη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. κηρύττω την έναρξη της συνεδρίασης. Πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η κοινή συζήτηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την πρόσβασή τους στα διαφθορτικά ταμεία και το θέμα του ορισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχουμε το Συμβούλιο και την Κομισιόν που θα κάνουν δηλώσεις για το θέμα της πρόσβασης στα διαφορετικά ταμεία και επίσης για την αξιολόγηση του ορισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εξ ονόματος του Συμβουλίου, ο κύριος Νικόλα Γουάμεν έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Θέλω να χαιρετήσω το γεγονό ότι το Κοινοβούλιο μα εστιάζει την προσοχή του στο θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Βρισκόμαστε σε ένα δύσκολο οικονομικό κλίμα και γι' αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι οι κύριοι συνεισφορείς στην οικονομική ανάπτυξη να έχουν ένα έφορο κλίμα μέσα στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν. Έχετε επιλέξει αυτή τη συζήτηση με δύο κύρια θέματα την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα διαρθωτικά ταμεία και τον ορισμό των, των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ήταν αυτά τα δύο τα αντικείμενα προφορικών ερωτήσεων προ το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Νομίζω ότι είναι σωστό να αντιμετωπίσουμε και τα δύο αυτά θέματα από κοινού. Είμαι σίγουρο ότι ο κύριο Επίτροπο θα μπορέσει να αντιμετωπίσει με πιο πολύ λεπτομέρεια τα συγκεκριμένα αυτά θέματα, τα οποία ενδιαφέρουν ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο σα, αλλά ενδιαφέρουν και την Κομισιόν. Από την πλευρά τη Προεδρίας θέλω να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες σκέψεις που είναι πολύ σημαντικές για το Συμβούλιο. Καταρχήν, οι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ο σκελετός της οικονομίας μας. Είναι η δημιουργή πλούτων. Είναι αυτή που μας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμοστούμε με ευέλικτο τρόπο σε αλλαγές σε ζήτηση και είναι η κύρια πηγή απασχόλησης. Γι' αυτό τον λόγο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 σε μια εποχή που έχουμε πάνω από 25 εκατομμύρια ανέργων, χρειαζόμαστε χρειαζόμαστε του, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης για τους νέους μας. Μέσα στο χρονικό διάστημα 2007 ως το 2014, τα διαρθρωτικά ταμεία έχουν δώσει περίπου 70 δισεκατομμύρια ευρώ στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Αυτή η οικονομική υποστήριξη βοηθά να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια τη Χρηματοπιστωτική κρίση και τη στενότητας πιστώσεων, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ακόμα πιο σημαντική. Γι' αυτό μια σειρά από προγράμματα εγγυήσεω δανείων προς τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν διευρυνθεί με πρωτοβουλίες που δίνουν <clears throat> επιδότηση επιτοκίων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επίσης για την βελτίωση της φεραγγιότητάς τους. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να δώσουμε μια υποστήριξη προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από τα διαρθρωτικά ταμεία. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εξασφαλίσουμε πιο αηφόρο ε, χρηματοδότηση αυτών των επιχειρήσεων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και στο μέλλον είναι απαραίτητο και το ίδιο κεφάλαιο καθώς και η δανειοδότηση για τις μικρομεσαίε επιχειρήσεις. Επιπλέον οι επιχειρήσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση σε δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με ευνοικού όρους. Και αυτό είναι ένα σημαντικός και πολύτιμο μηχανισμός χρηματοδότηση που δίνει εναλλακτικέ δυνατότητε από την δανειοδότηση μόνο και μόνο από εμπορικέ τράπεζε. Μία σημαντική επίσης πηγή χρηματοδότησης προέρχεται από τις κοινέ πρωτοβουλίες της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ο Τζέρεμι, η Τζέσικαν και ο Τζάνσον είναι εργαλεία που έχουν σαν στόχο να βελτιώσουν την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την παροχή μετοχικού κεφαλαίου, δανείων και εγγύησεων. Σε ό,τι αφορά τώρα τον ορισμό του τι αποτελεί μικρομεσαία επιχείρηση, η Κομισιόν κάνει μια ε, έρευνα για να δει ποιε είναι οι κατευθύνσει των κρατών μελών σε σχέση με αυτόν τον ορισμό και το αν είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί ο ορισμό αυτό. Το Συμβούλιο δεν έχει ακόμα ευκαιρία να συζητήσει για το θέμα αυτό και προσβλέπουμε στο να δούμε τι προτάσει τη Κομισιόν του του Λεχθέντο. Είναι σημαντικό να τονίσω ότι ο τωρινό ορισμό κάνει 95% όλων των επιχειρήσεων στην Ευρώπη να είναι μικρομεσαίες. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να έχουμε μια πλήρη συζήτηση για το τι ακριβώς είναι αυτός ο, ο καλύτερος, ο πιο πρόσφορος ορισμός. Περιμένω λοιπόν να ακούσω και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την άποψή σας. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κύριε Επίτροπε, το θέμα ενδιαφέροντά σα σήμερα, σήμερα το πρωί είναι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κάτι που είναι ζωτικό στο τωρινό οικονομικό κλίμα. Θα ήθελα να περατώσω την ομιλία μου τονίζοντα ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι μεν πάρα πολύ σημαντική, αλλά χρειάζονται και ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό κλίμα οι μικρομεσαίες επιχειρήσει για να μπορέσουν να ευδοκιμήσουν. Η νομοθεσία για τις μικρές επιχειρήσεις του 2008 ήταν πάρα πολύ σημαντική για τη δημιουργία ενός πλήρους πλαισίου του επιχειρήν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον πολλά κράτη-μέλη έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες με τη δημιουργία μόνο απευθυντικών θηρίδων για να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει όμως όλοι μας να παραμείνουμε επάγρυπνοι για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε πάντα το κατάλληλο περιβάλλον στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν και να απλοποιήσουμε τους κανόνες τους οποίους υπόκειται, να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και το διοικητικό άρθρο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Äh, Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, Κυρίε και κύριοι, οι επιχειρήσεις επιχειρήσει είναι ο πυρήνας η καρδιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. 23 περίπου εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουμε στην Ευρώπη. Είναι 99,8% των Ευρωπαίων επιχειρηματιών. Ανάπτυξη λοιπόν και μελλοντική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης που εξαρτώνται από την ανταγωνιστικότητα ακριβώς των μικρομεσαίων μας επιχειρήσεων. Η κρίση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ακριβώς όπως και όλες τις άλλες επιχειρήσεις τις έπληξε εξίσου και κατά κανόνα είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες τώρα που αντιμετωπίζουν για να εξεύρουν νέα κεφάλαια. Υπάρχει λοιπόν κοινή και δημόσια ευθύνη να βοηθήσουμε τις ΜΜΕ να μην γίνουν τα θύματα των πιστωτών τους αλλά με καινο, τόμα δράση να μπορέσουν να υλοποιήσουν το μεγάλο δυναμικό τους. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια επανειλημμένα ανέλαβε μέτρα ώστε η πρόσβαση αυτή των ΜΜΕ σε κεφάλαια να διευκολυνθεί και να βελτιωθεί. Μέσω της προσαρμογής υφισταμένων προγραμμάτων 2010 <clears throat> και 2011 καταφέραμε τα διαθέσιμα κεφάλαια και τα μέσα, τα χρηματοδοτικά μέσα για την εγγύηση δανείων να φτάσουμε σε πάνω από 1,8 δις ευρώ κατά το τέλος δηλαδή του 2010 και να αυξηθεί αυτό το ποσό. Έχουμε πολλά μέσα που χρηματοδοτήθηκαν από τα κράτη-μέλη. Πάνω από 90.000 θέσεις απασχόλησης άμεσα δημιουργήθηκαν με αυτά τα μέτρα. Θέλω να δραχθώ της ευκαιρίας εδώ και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ευχαριστήσω για την ταχεία υποστήριξη που δόθηκε στην τροποποίηση και προσαρμογή των κανονισμών μας που κατά τη διάρκεια των ετών κατέστησαν αναγκαία κατέστη αυτή η προσαρμογή για να αντιδράσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά στο πεδίο για παράδειγμα των ανακυκλούμενων δανείων ώστε να δραστηριοποιηθούμε και να πετύχουμε μια σημαντική συνεισφορά για την υπέρβαση της κρίσης ιδιαίτερα σε κάποια κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις. Κατά τα τέλη αυτού του έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκοινούμε τα κράτη-μέλη ανέλαβε περαιτέρω δράση ώστε να προσαρμοστούν με τέτοιο τρόπο τα προγράμματα ώστε τα ακόμα διαθέσιμα μέσα να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά στοχοθετημένα για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης αλλά επίσης και για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων που ήταν και αυτό θέμα αυτής της πρωτοβουλίας που αναλάβαμε. Πρόκειται λοιπόν ακριβώς ε, για αυτήν την ανακατανομή που εφόσον επιτρέπεται και από τα άλλα κονδύλια να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ωφεληθούν από αυτά διότι εκείνε είναι που δημιουργούν σε αηφορία, σε μακροπρόθεσμη συνιστόσα θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Να το υπενθυμίσω αυτό. Έχουμε 24 εκατομμύρια περίπου ανέργους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 23 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ας πούμε απλουστευμένα, αν κάθε μικρομεσαία επιχείρηση προσλάμβανε έναν άνεργο, θα είχαμε σχεδόν εξαλείψει το πρόβλημα της ανεργίας στην Ευρώπη αν γινόταν κάτι τέτοιο. Με βάση αυτή λοιπόν την πρωτοβουλία θα καταλήξουμε σε μια ανακατανομή υπό το σημερινό πρίσμα 5-8 δις ευρώ. Για την επόμενη προγραμματική περίοδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει σαφώς κέντρο βάρους υπέρ των ΜΜΕ, 80% των μέσων των κονδυλίων για τις ε, καλύτερα ανεπτυγμένες αλλά και τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές από άλλη δράση θα ωφελήσουν αυτές τις περιφέρειες ώστε μη με έψιλον στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην βελτίωση της αποδοτικότητας της εκμετάλλευσης ενέργειας να μπορέσουν να ωφεληθούν. Μην ξεχνάμε ότι σε απόλυτα μεγέθη είναι περισσότερο από 80% οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε τέτοιες περιφέρειες. Είναι ένα σαφές μήνυμα που στέλνουμε με αυτόν τον τρόπο ότι πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση των ΜΜΕ. Για να γίνει αυτό πρέπει από κοινού να συνεργαστούμε. Να υπάρξει η ρύθμιση της πρόσβασης σε τέτοια κονδύλια, σε τέτοια δάνεια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις πολλές προτάσεις για την διοικητική ανακούφιση και διευκόλυνση. Ταυτόχρονα υπενθυμίζω ότι ένα σημαντικό μέρος αυτών των μέτρων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο <clears throat> για παράδειγμα η υλοποίηση του Small Business Act που θα πρέπει και σε, να ε, προχωρήσει σε μια προϋπόθεση που θα λειτουργεί πάντα ε, αυτόματα. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Μια προσπάθεια χρειάζεται στο ευρωπαϊκό επίπεδο και στα κράτη-μέλη προς όφελος των ΜΜΕ. Ολοκληρώνω και καταλήγω σε ένα τελευταίο σημείο, το οποίο ήδη εθίγει πιο πριν. Ο ορισμός των ΜΜΕ. Πάντα δημιουργεί αυτό αφορμή για συζητήσεις. Γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτόν τον ορισμό σε τακτά διαστήματα τον επανεξετάζει και έτσι θα έχουμε μια περαιτέρω ανεξάρτητη αξιολόγηση που βρίσκεται υπό εξέλιξη, ώστε να δούμε τι θα πρέπει να γίνει σε σχέση με τα κονδύλια και τις δράσεις. Αναμένουμε το αποτέλεσμα αυτών των, ε, αυτής της μελέτης κατά την αρχή του, ε, της άνοιξης του 2013 ε, και θα πρέπει να δούμε αν θα καταλήξουμε σε μια αλλαγή του σημερινού ορισμού ή όχι. Κυρίες και κύριοι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. οικονομίας. Τους ε, τελευταίους μήνες και εβδομάδες μιλήσαμε πολύ για ανάπτυξη και όθηση προς την ανάπτυξη. Είναι σαφές, όποιος θέλει να δώσει τέτοια όθηση στην ανάπτυξη πρέπει να ξεκινήσει με τις ΜΜΕ, να ξεκινήσει με την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. Εμείς από πλευρά τη Επιτροπής είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Τώρα θα δώσω το λόγο στους ομιλητές ονόματος των πολιτικών ομάδων. Καταρχήν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, <clears throat> ο κύριος Μπέντσεν. E Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνουν πιο φιλικά για του ε, καταναλωτέ. Συχνά δυστυχώ συμβαίνει. Συμβαίνει το ότι αυτά τα προγράμματα από υπαλλήλου ε, για υπαλλήλου διατυπώνονται και όχι για του υπεύθυνου στην οικονομία. Και γνωρίζουμε όλοι ότι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει δημιουργούν θέσει απασχόληση. Και γι' αυτό θα έπρεπε εμεί εδώ τι διαδικασίε υποβολή αιτήσεων να τι καταστήσουμε πιο απλέ ε, και να τερματιστεί η γραφειοκρατία, η γραφειοκρατική επιβάρυνση Πρέπει να υπάρχουν και σαφέστερες ε, διασυνδέσεις ε, στην πρόσβαση για την ε, χρηματοδότηση επιχειρήσεων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε και πρέπει να αντιμετωπιστούν στην Ευρώπη. Έχουμε τέτοιες προκλήσεις και πρέπει να προχωρήσουμε για την αποδοτικότητα της ενέργειας. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα κομβικό σημείο για τη δυνατότητα χρηματοδότησης επιχειρήσεων και των προκλήσεων και στόχων που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Θα μπορούσαν από τα διαθροτικά κονδύλια να χρησιμοποιηθούν κονδύλια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να δημιουργήσουμε πολλές ευκαιρίες. Οι χειρόνακτες, οι εργαζόμενοι, οι εργάτες που εργάζονται εκεί θα μπορούσαν να συμμετάσχουν. Προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο, για τις κλιματικές αλλαγές, για την κλιματική προσαρμογή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ώστε οι ΜΜΕ να υποφεληθούν. Ακριβώς αυτές που δημιουργούν τις θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Ή ε, με αυτά τα επιχειρήματα θα έπρεπε να αναφέρουμε και δύο λόγια για τον ορισμό των ΜΜΕ. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ο ορισμό που υπάρχει να μην τροποποιηθεί υπερβολικά. Και θα έλεγα ότι αυτό θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη ακριβώς ότι μια και σήμερα 95% των επιχειρήσεων θα πρέπει να καλύπτονται. Γι' αυτό να μην έχουμε μεγάλες αλλαγές. Ευχαριστώ. Κυρία και τώρα... Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι. Τόσο συχνά και τόσες πολλές φορές αναφέρθηκε ότι η ΜΜΕ είναι η καρδιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και είναι η καρδιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και κάνουμε πολλά για αυτές. Αλλά είναι κάτι ξεχωριστό, διότι σε αντίθεση με άλλους μεγάλους οικονομικούς ε, εμπλεκόμενους έχουμε εδώ μικρές επιχειρήσεις που είναι ανταγωνιστικές και πρέπει να είναι ανταγωνιστικές στην παγκόσμια οικονομία και πρέπει να μπορούν να προσαρμόζονται στις νέες προϋποθέσεις και όρους. Αυτό είναι το ξεχωριστό των ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή και τις υποστηρίζουμε. Δεν θα ε, προωθηθούν στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο, αλλά γίνεται αυτό ήδη από σήμερα υπέρ εκείνων των επιχειρήσεων. Πολλά λοιπόν και για τα ε, κονδύλια και ε, για τα διαθροτικά κονδύλια γίνονται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να βελτιώσουν τα πράγματα αυτές οι δράσεις και να πλουστεύσουν τα πράγματα. Όταν μια μικρή επιχείρηση παίρνει ένα δάνειο και θέλει να ζητήσει με χαμηλό επιτόκιο τέτοιο δάνειο πρέπει να διευκολύνεται γραφειοκρατικά και να μην επιβαρύνεται. Να βελτιώσουμε λοιπόν τα πράγματα. Πιστεύω επίση ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσει με τη βοήθεια μια ευφυού και εφάνταση ε, δημιουργική προσέγγιση θα μπορέσουν να επωφεληθούν ώστε να συνδεθούν για την οικονομία, την ανάπτυξη, την ε, νέα πρωτοβουλία για την δημιουργία θέσεων απασχόληση. Ο επίτροπο Χάν σε μία από τι προηγούμενε συζητήσει το είχε πει αν κάθε μικρομεσαίο επιχείρηση προσλάμβανε έναν νέο άνεργο, τότε θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη. Δεν θα είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Έχει δίκιο με αυτό. Και θα πρέπει εδώ να εμείνουμε και να επιμείνουμε κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διατίθενται όταν απασχολούνται ένας ή δύο νέοι σε αυτές τις επιχειρήσεις. Θα μου θύμιζε κάτι τέτοιο το παρελθόν σε σχέση με τη λακροατική Γερμανία, όμως ένα εφάνταστο πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει πραγματικά αυθεντικές θέσεις κατάρτισης και απασχόλησης για τους νέους θα έδινε δυνατότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξίζει λοιπόν τον κόπο να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να πετύχουμε να λειτουργήσει ένα τέτοιο σχέδιο. Ίσως θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε μέχρι την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο να ευδοκιμήσουν τέτοιες ιδέες για τέτοια προγράμματα. Θα ήθελα να πω, δεν θέλω μόνο να έχουμε αυτές τις θετικές επιπτώσεις προσωρινά για αυτές τις επιχειρήσεις. Πρέπει μακροπρόθεσμα σε ένα χρονορίζοντα να υπάρξουν θετικά ε, αποτελέσματα, ωφέλη. Ένα πράγμα ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρω ότι υπάρχει αναδιατύπωση του δικαίου για τον ανταγωνισμό. Θα θέλαμε σε σχέση με τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην ισχύουν απόλυτα διαφορετικοί όροι και προϋποθέσεις. Και αυτό δημιουργεί γραφειοκρατική επιβάρυνση και δυσχεραίνει την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Πρέπει να υποβάλει θετικέ προτάσει για τι περιφέρειε. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Για τους φιλελεύθερους ο κύριος Κρόιτσμαν. Ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η πρόσβαση στα κονδύλια για τα δάνεια και πιστώσεις. Η πολιτική συνοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει εδώ. Υπάρχουν διαφορετικά προγράμματα, ήδη προαναφέρθηκαν. Μία μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τι επιπτώσει τη αποτελεσματικότητα τη διάθεση κονδυλίων των διαθροτικών ε, ταμείων και άλλων κονδυλίων που στοχεύουν στι ΜΜΕ απεκάλυψε τι ελλείψει. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των διαφορετικών τύπων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μικροεπιχειρήσει ε, ή οι ανεξάρτητοι επιχειρηματίε ε, που δεν έχουν πολλά, δεν έχουν ε, απασχολούμενους στην επιχείρησή τους. Έτσι λοιπόν η χρηματοδότηση προγραμμάτων και προχρηματοδότηση απαιτεί διαφοροποίηση των κανόνων και ρυθμίσεων για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Αυτό με οδηγεί στο να εκφράσω κάποιες παρακλήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να το καταφέρουμε για την πρόσβαση από τα διαθετικά ταμεία να διευκολύνουμε την πρόσβαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χρειάζεται βελτίωση και για την ε, ε, κατανομή των κεφαλίων. Χρειάζεται χρειάζεται μια πιο χαλαρή προσέγγιση για την προχρηματοδότηση προγραμμάτων και σχεδίων. Μια πιο στοχοθετημένη διαμόρφωση των κονδυλίων και τη διάθεση αυτών των κονδυλίων σε σχέση με τις διαφορετικές μορφές τέτοιων επιχειρήσεων. Μια διαφορετική διαμόρφωση των συγχρηματοδοτήσεων και σε σχέση με τον κύκλο απόσβεσης πάλι να λαμβάνονται αυτά τα στοιχεία που διαφοροποιούν μεταξύ τους τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπόψη. Εδώ τα επιμελητήρια μπορούν να δώσουν μια συνεισφορά εμπορικά και άλλα επιμελητήρια. Πρέπει να ενισχυθεί η διαμόρφωση ιδίων κεφαλαίων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να μπορούν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να παίρνουν τέτοια δάνεια. Είναι πολύ σημαντικό η Συμφωνία Βασιλεία 3 να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δυσχεραίνεται η χρηματοδότηση με δάνεια των ΜΜΕ, αλλά να δημιουργηθεί δυνατότητα χωρί τριβέ και προβλήματα, αν γίνεται, και πάντα με θετικού όρου να μπορούν να υποφελούνται οι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ευχαριστούμε. Τώρα για τους πράσινους η κυρία Μιράντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν Ο ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίε διαχειρίζονται πολλέ θέσει εργασία, παίζουν σημαντικό ρόλο σε περιοχέ όπου υπάρχει πρόβλημα στην απασχόληση των νέων, των γυναικών, των μεταναστών. Σε αυτή τη στιγμή σε πολλά κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν αυτές οι ομάδες του πληθυσμού μια ανεργία 50, ακόμα και 40, 50% ανεργίας. Όταν υπάρχει τόσο μεγάλη ανεργία πρέπει η πολιτική και όλοι μας να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα του οικονομικού αυτού τομέα στην Ευρώπη. Μικρές και, μεγάλες, και μεσές επιχειρήσεις με έχουν ε, υπερχρεωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια. 85% όλων των θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δημιουργηθεί από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδίως από νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θεωρούμε ότι είναι υπερβολικό το διοικητικό άκτο που πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτές οι επιχειρήσεις. Είναι απαραίτητο λοιπόν στην επόμενη μεταρρύθμιση των διαφορετικών πόρων να υπάρξει και ε, μια σειρά από νέα προγράμματα τα οποία θα κατευθύνονται ιδιαίτερα στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό θα ευκαμπτοποιήσουμε τους μηχανισμούς διοικητικής διαχείρισης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με καινοτόμα μέτρα, με πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες ή ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε πλήρως το δυναμικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να υπάρξει ευνόηση της δραστηριότητας σε διαμεθοριακό ε, επίπεδο και να μπορέσει να αντιμετωπιστεί καλύτερη κρίση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τώρα ο κύριος Τσίτσεστερ για την ομάδα του. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. το θέμα προβλέπεται μεν, αλλά δεν νομίζω ότι θα ακούσουμε πολύ ικανοποιητικέ απαντήσεις, γιατί το πρόβλημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν είναι μόνο πώς θα αρχίσουν τη δραστηριότητά τους, αλλά και πώς θα επιβιώσουν και πρέπει να τις βοηθήσουμε όσο μπορούμε, όσο λογικότερα γίνεται. Οι ανησυχίες τους είναι γνωστές εδώ και χρόνια. Πρώτον, χρειάζονται πρόσβαση σε πληροφόρηση βοήθεια για να μάθουν πού να απευθυνθούν. Δεύτερον, πρέπει να έχουν πρόσβαση και σε χρηματοδότηση. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να πάρουν μικρά δάνεια. Οι τράπεζες ε, θέλουν συνήθως να δίνουν πολύ ψηλότερα δάνεια για να έχουν υψηλότερα κέρδη και κάτι για το οποίο μπορούμε και εμείς κάτι να κάνουμε είναι να διευκολυνθεί η γραφειοκρατία που αντιμετωπίζουν. Είναι πολύ δύσκολο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις να την αντιμετωπίσουν, δυσκολότερο από ό,τι στις μεγαλύτερες. Και τέλος, μακροπρόθεσμα ελπίζω η Κομισιόν να καταλάβει και το τελευταίο σημείο της ερώτησής μας για την χρήση ποσών που δεν έχουν διατεθεί για να βοηθήσει από άλλες θέσεις του προϋπολογισμού τη μικρομεσές επιχείρηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Αλαβράκος για την ομάδα του. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής οικονομίας και αποτελούν ίσως το πιο σημαντικό εργαλείο για την τόνωση της ανάπτυξης και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης υπό τα σπαρούσα συνθήκας που κυριαρχούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, ο κλάδος είναι ο πλέον ευάλωτος στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης η μείωση της κερδοφορίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ελλάδα φτάνει το 60% και αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό στην ευρώπη ενώ ακολουθεί η ισπανία με ποσοστό 55%. στον αντίποδα βρίσκεται η γερμανία που καταγράφει εκτείναξη της κερδοφορίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ποσοστό 21%. στην πατρίδα μου την ελλάδα παρατηρείται η μεγαλύτερη επιδείνωση στον κλάδο και η δυνατότητα πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηματοδότηση είναι πλέον ανύπαρκτος. πολλές επιχειρήσεις κλείνουν με αποτέλεσμα την επιδείνωση της επιχειρηματικότητας και της εργασίας. ωστόσο τελευταίες έρευνες της ευρωπαϊκής τράπεζας που αφορούν τις δανειοδοτήσεις δείχνουν ότι έχουν αυξηθεί τα κριτήρια από τις τράπεζες για την χορήγηση δανείων στι μικρομεσαίες. καλείται λοιπόν η επιτροπή να μελετήσει και να προτείνει μέτρα για τη διευκόλυνση της απορροφικότητας των κονδυλίων στις χώρες κυρίως που αδυνατούν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα ποσά συγχρηματοδότησης λόγω αυστηρών προγραμμάτων λιτότητος. Να προωθήσει συνεργασίες και συνέργειες μεταξύ του Διορθωτικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ώστε να βρεθούν χρηματοπιστωτικά εργαλεία και να μπορούν να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Να βρεθούν οι πιο κερδοφόροι τομείς σε κάθε οικονομία και να γίνει ένας σωστός στρατηγικός προσανατολισμός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλά μπορούν να αναφερθούν για την ανάγκη να αναπτύξουμε μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολλά μπορούν, πολλά μπορούν να αναφερθούν γιατί για το πόσο είναι σημαντικέ οι ΜΜΕ για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Μπορεί κανείς να αναφέρει πολλά. Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι η εφαρμογή αυτών των μέτρων λιτότητας οδηγούν αυτά τα μέτρα κάθε μέρα στο να στραγγαλίζονται πάμπολες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αν δεν υπάρξει ρήξη όσον αφορά τις ε, πολιτικές λιτότητας ε, και αν δεν υπάρξει προώθηση πραγματικής οικονομικής ανάπτυξης δεν θα γίνει τίποτα. Έχουμε εδώ την ε, λιτότητα που δημιουργούν μια υπέρβαση σε σχέση με αυτή την οδηγία. Δεν δημιουργούμε παρά μόνο αυταπάτες για το κρύβονται πολλά πίσω από ωραία λόγια χωρίς να υπάρχουν αποτελέσματα και έχουμε δραματικές επιπτώσεις που επομίζονται όλοι. Γι' αυτό τα μέτρα που έχουν ε, επιβληθεί από την Τρόικα στην Πορτογαλία είναι ένα καλό παράδειγμα αυτής της δραματικής κατάστασης. Ε, καταστράφηκαν στην Πορτογαλία 200 ε, τόσες χιλιάδες θέσεις απασχόλησης. Έχουν καταστραφεί και καταστρέφονται καθημερινά θέσεις απασχόλησης. Πολλοί από αυτούς τους απασχολούμενους που καταστράφηκαν οι θέσεις απασχόλησής τους είναι εργαζόμενοι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει κάτι να γίνει. Εδώ έχουμε περί περικοπές μισθολογικές και έχουμε και φορολόγηση όσον αφορά τα προϊόντα που πολλούνται από αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που οδηγούν μετά σε προβλήματα όσον αφορά και την κατανάλωση και δημιουργούνται πάμπολα προβλήματα εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρέπει εδώ τα μέτρα αυτά τα οποία έχουν ιδιαίτερα πλήττουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντιμετωπιστούν. Γίνεται σήμερα λόγος για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι σημαντική αυτή η πτυχή, αλλά θα πρέπει πρέπει να μην εφαρμόζονται πολιτικά μέτρα που ακριβώς καταδικάζουν ε, μέσα σε αυτή τη συγκυρία τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στο να μην μπορούν ε, να επιβιώσουν. Πρέπει επίσης και η δημόσια υποστήριξη και ο μονοπωλιακός χαρακτήρας που δημιουργείται και με την, το μεγάλο κεφάλαιο που υποφελείται και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πρέπει να μπορέσουμε να δράσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχουμε έχουν ε, την ε, ε, κατάσταση μονοπωλιακών τιμών που επιβάλλονται σε αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τους ανταγωνιστές. Πρέπει να διευκολύνουμε την γραφειοκρατική επιβάρυνση, να ανακουφίσουμε την κατάσταση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για εκείνους ιδιαίτερα που αντιμετωπίζουν αυτές τις μεγάλες δυσκολίες. Ευχαριστώ. Και τώρα στη συνέχεια, λίγο προεδρεύον, θα προχωρήσουμε με την κυρία Σίνκλερ. Ένα μισή λεπτό παρακαλώ. Συγγνώμη, συγγνώμη λέει κυρία ε? Σίνκλερ. Πολύ ωραία είναι αυτά τα λόγια που ακούσαμε σήμερα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει που είναι η ραχοκοκαλιά τη οικονομία και τη κοινωνία τη Ευρώπη. Μα είναι κοντά στην πραγματικότητα όλα αυτά. Μας ε, έχουν πει κάποτε ότι ήμασταν το Ηνωμένο Βασίλειο ένα κράτος μαγαζατόρων. Αλλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες έχουν τις περισσότερες επιχειρήσεις. Εγώ βλέπω κάθε φορά στην εκλογική μου περιφέρεια να μου λένε αυτοί που έχουν μικρά μαγαζιά ότι μας στραγγαλίζουν οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει πρόσβαση σε κονδύλια, δεν υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος καθαρός νησφορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν παίρνει αρκετή βοήθεια, δεν παίρνει την απαραίτητη εκπαίδευση που χρειάζεται. Όλες οι άλλες ε, ε χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πρόσβαση στα κοινοτικά ταμεία καλύτερη από αυτήν του Ηνωμένου Βασιλείου. Στις ε, αγγλικές επιχειρήσεις λοιπόν δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Όλη η χρηματοδότηση του Τζέρεμι που είναι μικρομεσές, υποστηρίζει τις μικρομεσές επιχειρήσεις, δίνει χρηματοδότηση στη Γαλλία αλλά τίποτα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό είναι έσχος. Και όπως σας είπα, είμαστε ο δεύτερο καθαρός συνεισφορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να σταματήσουμε τους ενδιάμεσους να χρηματοδοτήσουμε κατευθείαν τις δικές μας μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σίνκλερ. Τώρα θα συνεχίσουμε με άλλους ομιλητές. Πρώτος ο κύριος Ρούμπικ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα μια ερώτηση προς τον Επίτροπο Χάν θα είχα. Και τι γίνεται σε σχέση με την ε, έρευνα για τις υποδομές και τι σχεδιάζεται σε σχέση με τις υποδομές για την έρευνα ιδιαίτερα ως μια προσφορά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προβλέπετε κάτι τέτοιο. Η δεύτερη ερώτηση είναι προς τον Υπουργό Βάνεν και από τον Πρωθυπουργό Προεδρεύον, Πρόεδρο Ολάντα ακούσαμε ότι χρειαζόμαστε τα κατεπηγόντας μια στρατηγική για την ανάπτυξη. Πώς αυτό θα έχει επιπτώσεις άμεσα στον προϋπολογισμό του 2013. Ποιες θέσεις και ποια κονδύλια στον προϋπολογισμό 2013 μπορούν να προβλεφθούν για μια συγκεκριμένη τέτοια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη που θα μπορούσε να δρομολογηθεί και τι μπορεί να γίνει σε σχέση με το ε, πρόγραμμα πλαίσιο μέχρι το 2020 ποιες δομές ε, για την ανάπτυξη προβλέπονται και ποια προγράμματα θέλετε να ωφεληθούν και κυρίως με ποια κονδύλια θα προοικοδοτηθούν. Τρίτη παρατήρηση. Πρέπει να μεριμνήσουμε οι νέε γυναίκε επιχειρηματίε ε, και οι νέοι επιχειρηματίε να έχουν ευκαιρίε στι άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να συλλέξουν τέτοιου είδους εμπειρία. Υπάρξουν, υπάρχουν τα προγράμματα Εράσμους για τους νέους επιχειρηματίες. Θα υπάρξει αύξηση κονδυλίων ώστε οι νέες γυναίκες επιχειρηματίες ε, να μπορέσουν ε, να έχουν πρόσβαση στις αγορές ε, και στους εμπλεκόμενους αυτές και να προβληματιστούμε επίσης για το πώς θα μπορέσουμε σε εκείνες τις επιχειρήσεις που έχουν ιδιαίτερο ρόλο στις εξαγωγές πώς μπορούμε να τις υποστηρίξουμε ίσως με το Ταμείο της παγκοσμιοποίηση και τα κονδύλια του. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε. Και τώρα για τρία λεπτά η κυρία Τόγια. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ανάπτυξη δεν είναι πολυτέλεια, είναι υποχρέωση. Όλοι αυτοί που γνωρίζουν το πόσο σημαντική είναι η οικονομική ανάπτυξη το έχουν καταλάβει αυτό. Η ομάδα μου έχει περηφάνεια για το γεγονός ότι πάντα έχει επιμείνει στην ανάγκη της ανάπτυξης, το οποίο σημαίνει πολλές φορές την ανάγκη διορθώσεων και ορισμένων ευρωπαϊκών πολιτικών. Όταν έχουμε λοιπόν προβλήματα με τις παραγωγικές δομές της Ευρώπης θα πρέπει να κάνουμε κατεπίγουσες αλλαγές. Χρειάζονται δράσεις οι οποίες να είναι πιο μακρόπνοες, οι οποίες να ασχολούνται με το ανθρώπινο κεφάλαιο, με τους νέους Ευρωπαίους και τις νέες Ευρωπαίες που θα πρέπει να εμφορούνται από ένα επιχειρηματικό πνεύμα να το κάνουν επιτυχία το να έχουν μια επιχείρηση γιατί αυτό βοηθάει και την οικονομία μας και την κοινωνία μας να υπάρχει λοιπόν διάχυτο επιχειρήν το οποίο θα οδηγήσει σε μια καλύτερη και πιο αηφόρο ανάπτυξη όπως ανέφερε και η κυρία Κρέλ γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε μια καινοτομία να χρησιμοποιήσουμε τις νέες ευκαιρίες αλλά συγχρόνως αυτό το επιχειρήν πρέπει να είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο μέσα σε αυτές τις μακρόπνοες δράσεις σκέφτομαι και το να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε και την ε, εκπαίδευση και την κατάρτιση. Έχουμε χάσει πάρα πολλά τεχνικά ιδρύματα στην Ευρώπη που δίνουν στους νέους τη δυνατότητα να καταλάβουν καλύτερα την ε, τεχνολογία και την επιστήμη και να τα χρησιμοποιήσουν στην καθημερινή του ζωή. Είναι απαραίτητο και το θέμα των πόρων για αυτή την πρωτοβουλία. Το λέω ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση της Κομισιόν. Φυσικά είναι το Συμβούλιο που θα αποφασίσει για τον κανονισμό των διαφθορτικών πόρων μαζί με το Κοινοβούλιο, αλλά είναι απαραίτητο να υπάρξει καλύτερο συντονισμό των πόρων που θα χρησιμοποιήσουμε τον τομέα αυτό. Θα πρέπει να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα διάφορα αυτά κονδύλια για την έρευνα, για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους διαφορετικούς πόρους, να υπάρξει μια συμπληρωματικότητα όλων αυτών των ε, ταμείων για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια σωστή λειτουργία. Αλλιώς θα έχουμε αλληλοεπικάλυψη και κατακαιρματισμό που θα είναι αρνητικό. Κάτι ακόμα θέλω να σας πω κύριε Επίτροπε, είναι σημαντική η εστίαση σε συγκεκριμένες κατηγορίες θεματικές, αλλά πρέπει να διατηρήσουμε και την περιφερειακή αυτονομία σε σχέση με την επιλογή των προγραμμάτων, γιατί ναι, υπάρχουν ορισμένε περιοχές οι οποίες έχουν την ανάγκη να έχουν μια βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το σχεδιασμό, αλλά υπάρχουν άλλες περιοχές που έχουν αυτόνομη ικανότητα να θεσπίσουν τα προγράμματα που θέλουν να ακολουθήσουν. Θα πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε τις περιφερειακές διαδικασίες που προωθούν το επιχειρήν τις θέσεις απασχόλησης και τις δυνατότητες να συνενώσουν όλους τους φορείς πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς σε ένα εδαφικό ε, επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να συνδυάσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική και την πολιτική των τοπικών αρχών. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει συντονισμό των δράσεων και των πόρων. Τέλος, για τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. <coughs> Πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να εμπλέξει όχι μόνο τα κράτη-μέλη, και όχι μόνο να λάβουμε υπόψη στοιχεία διαρθρωτικά όπω είναι η απασχόληση, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και ποιοτικά στοιχεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο σε μια περιφέρεια, αλλά έχουν στραμμένο το βλέμμα του προ όλο τον κόσμο. Όχι μόνο λοιπόν το τι κάνουν σε αυτή την περιοχή, αλλά τα δίκτυα μέσα στα οποία εμπλέκονται αυτέ οι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Μανέσκου για δύο λεπτά. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κύριε Επίτροπε. Η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε κονδύλια είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Είναι μεγάλη ευρωπαϊκή και εθνική πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Οι ΜΜΕ πλήττονται ιδιαίτερα από την σημερινή οικονομική κρίση τα κονδύλια των διαθροτικών ταμείων είναι μια μεγάλη ευκαιρία ώστε να επιτραπεί να επιβιώσουν με την ενίσχυση αυτών των κονδυλίων οι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Ο ρόλο τη ΕΕ και των εθνικών κυβερνήσεων έχει τεράστια σημασία όταν πρέπει να και πρόκειται να ληφθούν μέτρα ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε δάνεια και πιστώσει των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να δρουν αποτελεσματικά. Και κάτι άλλο το ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο ρυθμίζει την πρόσβαση των ΜΜΕ σε τέτοιες ε, δυνατότητες είναι υπερβολικά επιβαρημένη υπόθεση top heavy. Αυτό οδηγεί στο να μπορούν να ποθαρινθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντί να ενθαρρυνθούν. Αν θέλουμε να έχουμε ένα υψηλό ποσοστό συμμετοχής ε, όσον αφορά τα κονδύλια των διαθετικών ταμείων για τον ιδιωτικό τομέα χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα απλούστευσης. Πρέπει να ανοίξουν, να αλλάξουν οι κανονισμοί και οι διατάξεις, να ξεφορτωθούμε την γραφειοκρατική επιβάρυνση, να βελτιώσουμε την κατάσταση και να βελτιωθεί η κατάσταση των επιχειρηματιών μας μας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τηρήσατε το χρονικό όριο. Τώρα ο κύριος Μπιουτικόφερ. Ένα λεπτό παρακαλώ. Μάικ, Μικρόφωνο παρακαλώ. Yeah. Οι αγαπητοί συνάδελφοι οι οποίοι έχουν ε, προκαλέσει αυτή τη συζήτηση με, το, με τα ερωτήματά τους έθεσαν το ερώτημα του αν είναι ορθό να υπάρχουν συγχρηματοδοτήσεις για προγράμματα τα οποία ε, αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αν θα πρέπει να αναθεωρηθεί αυτή η διαδικασία. Αυτό είναι ένα σωστό θέμα, αλλά θα πρέπει να δούμε καλύτερα και το πλαίσιο μέσα στο οποίο εγγράφεται αυτό το ερώτημα και αυτή η προβληματική. Όταν εμείς έχουμε ένα ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που τον διευρύνουμε, τότε θα μείνουν πολύ λιγότερα κονδύλια για να διανεμηθούν σε αυτές που μέχρι στιγμής καλυπτόντουσαν ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γνωρίζουμε ότι τα οικονομικά μέσα δεν είναι επαρκή δεύτερον. Αν μειώσουμε τις προϋποθέσεις για συγχρηματοδότηση, τότε πάλι θα σημαίνει αυτό ότι είναι πολύ λιγότερες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε αυτό το πλαίσιο χρηματοδότησης. Επομένως, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε τέτοια διεύρυνση των ορισμών μόνο όταν έχουμε περισσότερα μέσα στη διάθεσή μα για να διανύμουμε στι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Δεν μπορούμε εμεί να φανταστούμε ότι μέσα στα πλαίσια του κόσμου και τη Ευρώπη 2020 να δίνονται στο μέλλον λιγότερα κονδύλια για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει από ό,τι τώρα. Κύριε Μπιτικόφερ, έχει τελειώσει ο χρόνο σα. Γι' αυτό σα αφαιρώ το λόγο, πρέπει να σεβόμαστε τον κανονισμό όλοι. Λοιπόν, Φόρντ, κυρία Βίκη Φόρντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι μικροεπιχειρήσεις πρέπει να εξαιρούνται από μεγάλα τμήματα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για να έχουν δικές τους διευκολύνσεις μεταξύ των οποίων και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Πολλές φορές μιλάμε για ποσά που θέλουμε να διαθέσουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά ακούω όλο και περισσότερα παράπονα από αυτές για το άχθος της γραφειοκαρατίας και πολλές φορές οι προβλεπόμενες πληρωμές δεν καταλήγουν ποτέ ενώ όποτε μία μικρή επιχείρηση έχει κάνει σωστά τη δουλειά της πρέπει και να πληρώνεται. Πολλές φορές δεν προσέχουμε τις επιπτώσεις και την εφαρμογή της νομοθεσίας που προβλέπουμε. Πρέπει να σταματήσουμε πλέον να μιλάμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να αρχίσουμε τη δράση. Εμείς θέσαμε εννέα συγκεκριμένα ερωτήματα και προσβλέπω σε εννέα συγκεκριμένες απαντήσεις κύριε Επιτροπέ μου. Μάλιστα. Και τώρα για ένα λεπτό ο κύριος Σιμάνσκι. Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατανοεί ότι η Κομισιόν θέλει να αρθούν οι φραγμοί στη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να διατεθούν περισσότερα κονδύλια σε αυτές. Στη χώρα μου διατίθενται αρκετά υψηλά κονδύλια για τις επιχειρήσεις, αλλά οι μικρομεσαίες δεν επωφελούνται επαρκώς, γιατί η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά. Η λογική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οδήγησε, μας δείχνει ότι είναι οι περισσότερες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα δύο τρίτα από αυτές είναι ανεξάρτητες άνθρωποι δηλαδή που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και για τους άλλους. Επίσης υπάρχει η κρίση λόγω της οποίας πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει συγχρηματοδότηση που να συμπεριλαμβάνει και τους ίδιους πόρους της επιχείρησης. Πρέπει το Κοινοβούλιο να απλοποιήσει τους κανόνες για τις πληρωμές αυτές. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Στογιανόφ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εδώ και πολλούς μήνες επισκέπτομαι τμήματα της Βουλγαρίας και έχω συνομιλήσει με πολλούς εκπροσώπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων που όλοι λένε το ίδιο. Μας πνίγουν προσέχετε μόνο τις τράπεζες και τις μεγάλες επιχειρήσεις ενώ εμείς πληγόμαστε χειρότερα από την κρίση. Δυστυχώς πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την απαρχαιωμένη τεχνολογία από την εποχή που άρχισαν την δραστηριότητά τους και χρειάζονται, τους ρώτησα, γιατί δεν ζητάτε ενωσιακά χρήματα για να εξυγχρονιστείτε και μας λένε πάντοτε ότι είναι πολύ μεγάλο το γραφειοκρατικό άχθος. Υπάρχει και ακόμη, ακόμη και η διαφθορά πλήττει ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί όλοι ενδιαφέρονται μόνο για μεγάλα και σημαντικά προγράμματα από μεγάλες επιχειρήσεις. Όσο για τους ορισμούς, να μην χρησιμοποιούμε τον αυστηρότερο, αλλά να, με έναν ευρύτερο ορισμό να τις βοηθήσουμε. Ο κύριος Φανίστερο, ένα λεπτό, ευχαριστώ. Θα πρέπει εδώ να υπάρξουν πιο θετικές προσεγγίσεις από τις τρινοδίες που ακούσαμε. Πιστεύω ότι με αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια από τα διαθετικά ταμεία και η κληρονομιά των επιχειρήσεων διατηρήθηκε και πολλές νέες επιχειρήσεις ε, μπόρεσαν ε, να αναδυθούν. Στην Ολλανδία, για παράδειγμα, 400 ε, έως χίλιες θέσεις απασχόλησης μπόρεσαν να διασφαλιστούν. Τα κεφάλαια που προσφέρονται πρέπει αποκεντρωμένα να μπορούν να δράσουν. Μέσα στο πλαίσιο 2014-2020 που συζητούμε σήμερα αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο δεν θα μπορούσαμε να προβληματιστούμε πώς θα μπορέσουν αυτά τα κονδύλια να διατεθούν επίτροπε. Έχουμε και το άτυπο Συμβούλιο Κορυφής, την Σύνοδο Κορυφής αύριο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι περισσότερο ώστε να επανεξετάσουμε αυτό το πλαίσιο πλαίσιο δεν θα μπορούσαν να απελευθερωθούν τέτοια κονδύλια, δεν θα μπορούσε κάθε χώρα να υποβάλει ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάποιες χώρες οι ίδιες δεν είναι καθόλου αθώες επειδή έχουν επιβαρύνει τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιδιαίτερα με το τη γραφειοκρατική επιβάρυνση. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά λοιπόν. Οι επιχειρήσεις ε, δεν μπορούν μόνες τους να κάνουν κάτι. Πρέπει να δώσουμε λοιπόν μια σημαντική προώθηση σε αυτά τα τρία θέματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για δύο λεπτά ο κύριος Κάρφιν παρακαλώ. Επίτροπε κύριε Υπουργέ, όλοι συζητούμε και λέμε ότι κάτι πρέπει να γίνει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να υπάρξει λιγότερη γραφειοκρατική επιβάρυνση, να υπάρξει μια καλύτερη πρόσβαση στις αγορές ε, για αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολλά κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πολύ περισσότερα, πολλά περισσότερα θα μπορούσαν να γίνουν. Πρώτον, πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Πιστεύω ότι σαφώς πρέπει να αυξηθούν οι δυνατότητες για προκαταβολές σε τέτοιες επιχειρήσεις, στις μικροεπιχειρήσεις και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Είναι πολύ δύσκολη η συγχρηματοδότηση ως πλαίσιο για αυτές τις επιχειρήσεις. Το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να επανεξεταστεί, πιστεύω. Είμαι εισηγητής για αυτό αυτό το θέμα. Επίσης, όσον αφορά και την συμμετοχή των διαθετικών ταμείων και την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρέπει εδώ να υπάρξει στις προηγμένες ε, τεχνολογίες δυνατότητα ε, πρόσβασης ε, για αυτές τις επιχειρήσεις. Συνολικά όλα αυτά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βελτίωση της κατάστασης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συγχρηματοδότηση εξετάζουμε κάτι που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιηθούν τα μη αντλημένα, μη χρησιμοποιηθέντα κονδύλια υπό αυτό το πλαίσιο όχι μόνο για την πρόθεση της απασχόλησης αλλά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ξεχωριστά. Αντιμετώπιση της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης. Όχι μόνο βέλτιστες προκτικές πρέπει να διαχέονται αλλά να υπάρχει και αντίστοιχη δράση όσον αφορά τα κράτη-μέλη διότι εδώ υπάρχει διαφορετική διαφορετική τοποθέτηση από τα κράτη-μέλη πολλές φορές και τρίτον να διευκολύνουμε την πρόσβαση στις αγορές. Αυτό πιστεύω είναι πολύ σημαντικό υπό τους όρους της διεύρυνσης της ψηφιακής αγοράς και των ευκαιριών που προσφέρονται με την ψηφιακή ημερήσια, το ψηφιακό θεματολόγιο και να δούμε και την δυνατότητα διεύρυνσης δυνατοτήτων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πολλές φορές δεν έχουν επαρκή πρόσβαση σε αυτές τις δυνατότητες. Σας ευχαριστούμε και για ένα λεπτό τώρα Hall. Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μεγάλα προβλήματα να εκμεταλλευτεί το Τζέρεμι. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ η εφαρμογή αυτού του μέτρου. Εμεί θα πρέπει να βοηθήσουμε τι μικρομεσαίες επιχειρήσει με το να ενσωματώσουμε στο, στην πολιτική για αυτέ τι εγγυήσει και τα μέτρα πρόθεση. Δεν υπάρχει μία μονάχα ε, λύση για την έλλειψη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στι πιστώσει. Η κυρία Μπάουλς προσπαθεί να επιφέρει κάποιε τροπολογίε στι οδηγίε για κεφαλουχική επάρχεια, αλλά χρειάζονται μικρομεσαίε επιχειρήσει και άλλου τρόπους χρηματοδότηση πέραν του τραπεζικού τομέα. Θα πρέπει να υπάρξει και μια αναλογικότητα σε σχέση με τα πρότυπα λογιστική και λογιστικού ελέγχου των επιχειρήσεων. Δεν έχει νόημα να έχουν δυνητικά χρηματοδότηση όταν έχουν τόσο πολύ γραφειοκρατία να υπερπηδήσουν που καμία μικρή επιχείρηση, μικρομεσαία επιχείρηση δεν μπορεί να δαπανίσει τον χρόνο να για πρόσβαση σε τέτοια χρηματοδότηση. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν διαφορετική βοήθεια σε όλε τι επιχειρήσει, ακόμα και τι μικρότερε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο Χρυσόγελο έχει το λόγο. Πράγματι η κρίση σήμερα πλήττει κυρίω τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και βλέπουμε να υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ανέργων που, είναι, που ήταν εργαζόμενοι σε τέτοιε επιχειρήσει, αλλά ταυτόχρονα και οι ιδιοκτήτες αυτών των επιχειρήσεων ε, χάνουν τη δουλειά τους και αυτό δεν καταγράφεται πολλές φορές στα ποστά ανεργίας. Σήμερα έχουμε ένα διπλό πρόβλημα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση αφενός σε δάνεια αλλά ούτε και σε χρηματοδοτήσεις από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι γεγονός ότι το 80% των αιτήσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων προ τι τράπεζε για δάνειο απορρίπτονται σήμερα στην ελλάδα άρα δεν υπάρχει χρηματοδότηση ούτε καν για να κινηθούν ούτε για να εισάγουν πρώτε ύλε ή προϊόντα άρα οδηγούνται σε κατάρρευση. Από την άλλη μεριά, οι όροι που εφαρμόζονται, που ισχύουν για την πρόσβαση σε ευρωπαϊκέ χρηματοδοτήσει, επίση δεν δίνουν τη δυνατότητα στι μικρομεσαίε επιχειρήσει να κινηθούν. Δηλαδή, πρέπει πρώτα να δαπανίσουν το κεφάλαιο, δεν είναι επιλέξιμο το ΦΠΑ και στο τέλο περιμένοντα μετά από πολύ καιρό να πάρουν πίσω τα χρήματα που έχουν δαπανήσει. είναι αδύνατο αυτό στην εποχή κατάρρευση. πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτό που είπε ο κύριο επίτροπο κάθε μικρομεσαία επιχείρηση να προσλάβει ένα νέο να συνδυάσουμε τι χρηματοδοτήσει για μικρομεσαίε επιχειρήσει με τι χρηματοδοτήσει για την αντιμετώπιση ανεργία των νέων για να μπορεί να γίνουν πράξει τέτοια. Ο Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι πάνω από 90% των επιχειρήσεων στην ΕΕ και δημιουργούν 80% των θέσεων απασχόλησης. Είναι η ραχοκοκαλιά λοιπόν της οικονομίας μας. Στην οικονομική κρίση ιδιαίτερα η πρόσβαση σε επαρκή κονδύλια δυσχεραίνεται για αυτές τις ΜΜΕ. Μία επίκαιρη μελέτη του Κοινοβουλίου καταδεικνύει ότι τα υφιστάμενα μέτρα ενίσχυσης δεν έχουν αρκετή το αποτέλεσμα και δεν είναι αρκετά στοχοθετημένα. Ο λόγος δεν διαφοροποιούνται μεταξύ των διαφορετικών ΜΜΕ και των χαρακτηριστικών τους. Δεν είναι μια ομοιογενής ομάδα όλη η ομάδα των ΜΜΕ. Εξαρτάται σε ποια, ακριβώς με ποια βάση και πώς δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Ένα νέο επιχειρηματίας που μόλι δημιουργεί τη δική του επιχείρηση είχε άλλε ανάγκε από μια παραδοσιακή κλασικού χαρακτήρα ε, μικρομεσαία επιχείρηση υπό οικογενειακή εκμετάλλευση. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν υπόψη αυτέ οι διαφοροποιήσει. Έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσει να μπορούν ανάλογα με τι ανάγκε του να αναπτυχθούν. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό τώρα η κυρία λουκατσέφσκα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι η βάση τη οικονομία μα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ανεργία και τη χρηματοπιστωτική κρίση. Είναι και η πηγή από την οποία παρέχεται απασχόληση και είναι φυσικά και μια πηγή οικονομική ανάπτυξη. 80% των νέων θέσεων εργασία, σύμφωνα με τι στατιστικέ, δημιουργούνται από μικρομεσαίε επιχειρήσει στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη 90% όλων των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες. Και επομένως είναι η βάση της απασχόλησης εκατομμυρίων ατόμων. Γι' αυτό όταν η Κομισιόν λέει ότι θέλει να αλλάξει τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει να λάβει υπόψη την, το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ελπίζω όταν κατανοήσετε ότι είναι νευραλικός αυτός ο τομέας για πάρα πολλούς εργαζομένους οι οποίοι θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη χρηματοδότηση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό ιδιαίτερα σε τομείς όπως είναι η επιστημονική έρευνα όπως είπε και ο κύριος Επίτροπος είναι η ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής ε, Οικονομίας και πρέπει να λειτουργεί καλά ο νιωτιαίος μυελός της Ευρώπης για να μπορέσει να λειτουργήσει και η υπόλοιπη Ευρώπη. Χρειάζεται λοιπόν καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, μείωση της γραφειοκρατίας, απλοποίηση των διακασιών που είναι τώρα ιδιαίτερα επαχθείς και χρονοβόρες. Και ο κύριος Επίτροπος θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα πρέπει να δώσουμε μία απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Γιατί μιλάμε για το πρόβλημα, δεν έχουμε απαντήσει ακόμα. Ευχαριστώ και τώρα ο κύριος Ντάρντεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι προφανές ότι η κρίση που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή πλήττει ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα πλαίσια της καταπολέμησης ιδίω της ανεργίας. Πολλοί συναδελφοί ζήτησαν απλοποίηση της ε, λειτουργίας των διαφορετικών ταμείων αλλά και στήριξη για την καλύτερη και ευκολότερη πρόσβαση σε αυτά. Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να διευκολυνθεί εδώ ο ορισμός της ΜΜΕ είναι σημαντικός. Ο ισχύων ορισμός αφορά πάνω από 67% των εργαζομένων στην Ένωση, σημαντικό μερίδιο δηλαδή της οικονομίας μας. Όπως συμβαίνει συχνά, πρέπει να βρεθεί και εδώ μια εξισορρόπηση ώστε το νομικό πλαίσιο να συνδυάζει και τον στόχο οικονομικής αποτελεσματικότητας και της σωστής προστασίας των εργαζομένων και του γενικού συμφέροντος. Μία ανισόρροπη μείωση των ε, βαρών που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ήταν όμως αρνητική. Παραδείγματος χάρη υπάρχει και το θέμα της ασφάλειας στην εργασία. Ιδίως για την προστασία της υγείας των εργαζομένων στους τόπους εργασίας. Η υγεία και η ασφάλεια δεν μπορούν να θεωρηθούν ως απλώς διοικητικά βάρη. Επίσης, η απλοποίηση των λογιστικών ορισμένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων τις ανησυχεί ιδιαίτερα, δικαίως νομίζω. Πώς θα μπορούσαν να παίζουν μεγαλύτερο ρόλο οι εργαζόμενοι και στη λήψη αποφάσεων για την επιχείρηση, αυτό εξαρτάται από τη δομή της λειτουργίας τους. Χρειάζεται ένα ελάχιστο όριο αδιαφάνειας. Και γι' αυτό αφού θέλουμε να μειωθούν τα βάρη της λειτουργίας τους δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποιος είναι ο στόχος της ύπαρξης αυτών των βαρών για να μην κάνουμε αδικίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πίπερ παρακαλώ ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάνουμε σήμερα λόγο για τα τα ταμεία για το πρόγραμμα ανάπτυξη, δηλαδή κυριολεκτικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στι πιο φτωχέ περιφέρειες. Δεν πρέπει να επινοήσουμε κάποια νέα ταμεία για την ανάπτυξη όπως κάποιες αριστερές κυβερνήσεις ζητούν στην Ευρώπη σήμερα. Εκείνα τα εκατομμύρια τα οποία σήμερα διατίθενται πρέπει στοχοθετημένα και γοργά να φτάσουν σε εκείνους που έχουν τις ανάγκες στις περιφέρειες έτσι η πρακτική εφαρμογή μπορεί να μας οδηγήσει να μάθουμε. Εκεί όπου ε, διαδικασίες για τον ανταγωνισμό υιοθετήθηκαν και ήταν υποχρεωτικές οι αιτήσει ε, για τη χρηματοδότηση, οδηγηθήκαμε στη δημιουργία πολυάριθμων επιχειρήσεων όπως ποτέ στο παρελθόν. Νανοτεχνολογίες, ε, τεχνολογίες εχμής σε συνδυασμό για την αποδοτικότητα στην χρήση ενέργειας, ενεργειακών πόρων, μπόρεσαν όλα αυτά βοηθήσουν αυτές τις επιχειρήσεις να στεφθεί με επιτυχία το εγχείρημά τους. Είναι αποτελεσματικές και είναι το αντίθετο ακριβώς στις αρχής της αδιάκριτης χρηματοδότησης χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Πρέπει να προχωρήσουμε έτσι. Στις μικρές επιχειρήσεις η υποστήριξη που δίνεται σε αυτές έχει σημαντική επίπτωση όσον αφορά την ανταγωνιστικότητά τους παγκόσμια. Αν το καταφέρουμε να είμαστε αποτελεσματικοί θα είμαστε αποτελεσματικοί και στην παγκόσμια με σκηνή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και 1,5 λεπτό τώρα ο κύριος Σβάμπ. Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μακρά παράδοση και αυτά τα οποία ακούσαμε σήμερα το πρωί στην συζήτηση στην Ολομέλεια δεν παρεκκλίνουν τόσο πολύ από αυτά τα οποία έχουν ακουστεί και στο παρελθόν ως προτάσεις. Πρέπει καταρχήν να πούμε προς την κυρία Βίκη Φόρντ ότι βέβαια δεν βοηθάει καθόλου να τον καταστήσουμε κάποιον υπεύθυνο γιατί τα πράγματα δεν ε, είχαν την τροπή που επιθυμούσαμε και την τελική έκβαση όπως το ευχόμαστε πρέπει εδώ να μην ε, ε, συνεχίσουμε την πορεία μας ε, αν αυτό δεν είναι επωφελές προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεύτερον, η στόχευση σε θέματα χρηματοδότησης δεν είναι τόσο επικοδομητική. Η αποκλειστική στόχευση σε αυτά τα θέματα. Εδώ βλέπουμε ότι στη Γερμανία δεν ενοχλούνται τόσο πολύ για τα θέματα χρηματοδότησης οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιμέρους αυτό μπορεί ίσως να είναι ένα πρόβλημα. Αλλά επειδή κυρίως το νομοθετικό πλαίσιο είναι τόσο περίπλοκο και δεδαλώδε που δεν μπορεί να είναι ένα διαφανέ πλαίσιο, αποτελεσματικό πλαίσιο για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Έτσι λοιπόν το θέμα του ορισμού που πρέπει να είναι πιο ακριβή και πιο στοχοθετημένο, πρέπει να είναι ένα σημαντικό μέσο όχι μόνο για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, αλλά και για την νομοθεσία γενικά σε αυτό το πλαίσιο. Και η έννοια που χρησιμοποιήσατε και είπατε ότι 99, τόσα τη είναι μικρομεσαίε επιχειρήσει, δείχνει δείχνει ότι υπάρχει συλλήβδη είναι ένα πρόβλημα επειδή δεν εξειδικευόμαστε και δεν διαφοροποιούμαστε σε σχέση με αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα καλύτερο ορισμό που θα είναι πιο αποτελεσματικός επιτέλους. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Δύο μπλε κάρτες για σας κύριε Σουάπ. Τις δέχεστε της κυρίας Βίκη Φόρτ πρώτα την μπλε κάρτα. Ευχαριστώ. Μια και αναφερθήκατε στη δική μου παρέμβαση, πρέπει να αποσαφηνίσω το τι συμβαίνει. Δεν κατηγορώ συλλήβδη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν διάφορε πτυχέ. Πρέπει να βρούμε συγκεκριμένε δεσμευτικέ λύσει όπου αυτό θα είναι δυνατόν. Εννέα συγκεκριμένα ζητήματα αναφέραμε και πρέπει να εξευρεθούν εννέα συγκεκριμένε απαντήσει για αυτά. Θα συμφωνούσατε μαζί μου ότι μια μικροεπιχείρηση που απασχολεί 5 έως 10 άτομα είναι πολύ διαφορετική από μια μεσαίου χαρακτήρα που απασχολεί απασχολεί περισσότερο, μέχρι 50 απασχολούμενους. Πρέπει λοιπόν να είμαστε διαφοροποιημένοι ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Η δεύτερη μπλε κάρτα είναι από την κυρία Σμιτ, παρακαλώ. Non, excusez-moi, c'était pour le catch the eye. Όχι, για τη διαδικασία catch the eye θέλω να λάβω το λόγο. Κύριε Σουάμπ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για το ερώτημα της κυρίας Φόρντ. Ακριβώς ακολουθεί την δική μου οδηγή γραμμή όπως και εσείς κυρία Φόρντ εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια να δώσουμε μια σαφέστερη έννοια στο τι σημαίνει μικρομεσαία επιχείρηση και να έχουμε κατηγορίε μέσα στι οποίε να θέτουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Όταν είναι πάνω από 90% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δεν μπορούμε να έχουμε μια στοχευμένη πολιτική. Επίση, υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι πιο μικρέ επιχειρήσει ενδιαφέρονται ιδιαίτερα στην έλλειψη γραφειοκρατία και στι απλοποιημένε διαδικασίε. Υπάρχουν όμω και μεσαίε επιχειρήσει στη δική μου ε, εκλογική περιφέρεια που είναι τόσο μεγάλε που να του ενδιαφέρει και ιδιαίτερα το θέμα τη χρηματοδότηση. Οπότε πρέπει να έχουμε διαφορετική στοχοδεσία για αυτέ τι επιχειρήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε και κύριοι. Ξεκινάμε την οφθαλμοσυλληπτική διαδικασία, αλλά έχω πάρα πολλού οι οποίοι έχουν ζητήσει το λόγο σε αυτή τη διαδικασία. Θα σας δώσω το λόγο, αλλά θα είμαι πάρα πολύ αυστηρός με το χρόνο. Ο κ. Κάλλιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα των μικρών μεσαίων επιχειρήσεων, γιατί αυτέ οι επιχειρήσει είναι η πιο σημαντική ομάδα επιχειρήσεων σε σχέση με τη δημιουργία θέσεων απασχόληση και για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την οικονομική κρίση. Να σταθούμε στον ορισμό των μικρών μεσαίων επιχειρήσεων. Όπως ελέγχθη, σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη εμπίπτουν σε αυτόν τον ορισμό, επομένως είναι ιδιαίτερα ασαφής αυτός ο ορισμός. Συμφωνώ με τη Βίκη Φόρντο ότι θα πρέπει να εστιάσουμε ιδιαίτερα στις μικρές επιχειρήσεις και στις μικρο, μικρού μεγέθους τέτοιε επιχειρήσει και να δώσουμε έμφαση στην αντιμετώπιση τη γραφειοκρατία και στην απλοποίηση των διαδικασιών. Δεν είναι μονάχα σημαντικέ από οικονομική έποψη, αλλά κοινωνικά Σημαντικέ Είναι αυτές οι οποίες κρατάνε ζωντανέ στις πόλεις μας. Χωρίς αυτές πεθαίνουν οι πόλεις μας. Να απαραίτητο λοιπόν να μειώσουμε τη γραφειοκρατία. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γία Κονσάρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το κλειδί εδώ είναι πώς θα βγούμε από την κρίση. Επίτροπε Χάν. Οι προοπτικές δεν είναι ρόδινες διότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα προσλάβουν κάθε μία από έναν εργαζόμενο αλλά μάλλον θα απολύσουν. Απαντού αυξάνεται το ΦΠΑ και αυτό είναι κακό για τις επιχειρήσεις υπηρεσιών γιατί αυξάνει τις τιμές μειώνονται οι μισθοί και οι συντάξεις και έτσι μειώνεται η ζήτηση. Για τον τομέα των υπηρεσιών λοιπόν κύριε Επίτροπε αυτά είναι πολύ άσκημα νέα. Η Επιτροπή πρέπει να μας βοηθήσει και τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν για αυτό το θέμα, αλλιώς όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ. Τρία θέματα πρέπει να υπάρξει καλύτερη και ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες αιτήσεων για χρηματοδότηση. Δεύτερον, δεν μιλήσαμε πολύ για την ανεπαρκή πληροφόρηση για δυνατότητες χρηματοδότησης για πρόσθετη χρηματοδότηση όπως από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή την ΕΤΕ. Και τρίτον, ερωτώ την Κομισιόν. Η συμμετοχή των ΜΜΕ στην εφαρμογή των μακροπεριφερειακών στόχων της Ένωσης πώς θα επιτευχθεί μέχρι στιγμής στη στρατηγική που αφορά την Βαλτική δεν έχω δει κανέ, ναι, καμία αναφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Τέλος, η Κομισιόν θα ενθαρρύνει τις χώρες μέλη να καταστρώσουν και εθνικά σχέδια στήριξης των ΜΜΕ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Βίνμπερν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έρχομαι από μία από τις φτωχότερες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βασίζεται ιδιαίτερα σε μικρές και μικροσκοπικές επιχειρήσεις. Παρά την ε, τροποποίηση των διαχρονικών πόρων, εμείς δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε μία αύξηση στο ΑΕΠ μας, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα τα ταμεία διαφορετικά για να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη. Όπως έλεγε, όπως ελέγχθη, αν κάθε μικρομεσαία επιχείρηση είχε τη δυνατότητα να απασχολήσει ένα άτομο παραπάνω, αυτό θα είχε μεγάλο αντίκτυπο σε οικονομικό επίπεδο και επίπεδο απασχόληση. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε τη δυνατότητα πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Όχι μόνο στην Τζέσικα και στον Τζέρεμι, αλλά γενικά. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει θα μα δώσουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Αν έχουν πρόσβαση σε διαρθρωτικά ταμεία θα μπορούν να τονώσουν ιδιαίτερα την οικονομία. Δεν θα πρέπει να θεωρούνται ότι είναι κρατικέ επιδοτήσει οι βοήθειε στις μικρομεσαίε επιχειρήσεις και να μην είναι αυτό πρόσχημα για τη μη χρηματοδότησή του. Ευχαριστώ. κύριος Κάρεντς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρώπη χρειάζεται ανάπτυξη. Για να μπορέσει να υπάρξει όμως οικονομική ανάπτυξη χρειαζόμαστε επενδύσεις. Μόνο με τις επενδύσεις θα μπορούμε να έχουμε νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε αυτή τη στιγμή περιορισμένους οικονομικούς πόρους που είναι στοχευμένοι ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι ιδιαίτερα ικανές στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Το πρόβλημα λοιπόν βρίσκεται στο γεγονός ότι ο ορισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι τόσο ευρύς αυτή τη στιγμή που περιλαμβάνει περίπου όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τουλάχιστον το 99% αυτών των επιχειρήσεων. Οπότε πολλές επιχειρήσεις που είναι πραγματικά μικρές, οι οποίες αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες, για να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση δεν έχουν ουσιαστικά τις ευκαιρίες που χρειάζονται. Θα πρότεινα να τροποποιήσουμε τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να περιλαμβάνει μόνο τις μικρές επιχειρήσεις που χρειάζονται τη μεγαλύτερη υποστήριξη. Ευχαριστώ. Η κυρία Τόια τώρα έχει το λόγο. Ο κύριος Σας ευχαριστώ πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι. Ξέρετε τον κύριο Χάμπτερμαν θα έπρεπε αν δεν τον ξέρετε να τον γνωρίσετε πριν από κάποιες δεκαετίες ε, ε, ίδρυσε μια επιχείρηση από το Πανεπιστήμιο Παντεμπορν. Σήμερα έχει εκατοντάδες εργαζόμενους ε, και για τα πήρε και το βραβείο το έπαθλο. Η κρατική υποστήριξη μπορεί να βοηθήσει. Τα κονδύλια αυτά μπορούν να βοηθήσουν τις μικρομεσίες επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε μια επιθετική προσέγγιση ίδρυσης νέων μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων. Πρέπει όμως να είναι χαμηλά τα κατόφλια, τα γραφειοκρατικά της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης χωρίς προβλήματα και προσκόμματα και πρέπει να υπάρξει ανακατανομή όσον αφορά τι δράσει για τη συνοχή. Για παράδειγμα, το τι πρέπει να γίνεται στην Ελλάδα για να μπορεί να παίρνει κάποια επιχείρηση κονδύλια. Χρειαζόμαστε και άλλε δράσει, ιδιαίτερα εκείνε που απουσιάζουν στι περιφέρειες. Είναι μια δυνατότητα αυτή. Χρειαζόμαστε και τι δύο λύσεις, και για τι περιοχέ τη περιφέρεια, αλλά και για καινοτόμε υψηλή τεχνολογία επιχειρήσει που θα τι βοηθούν αυτή είναι η επιταγή που πρέπει τώρα να εξαργυρώσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα στη συνέχεια κυρία Κάρπατς παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Οι μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις λοιπόν αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα διότι δεν έχουν πρόσβαση στα κονδύλια που χρειάζονται. Και αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Σημαντικότατη πρόκληση. Σε αυτόν τον το, τομέα πρέπει τα κονδύλια των διαθροτικών ταμείων να τα χρησιμοποιούμε καλύτερα. Πρέπει να επιταχυνθούν οι ρυθμοί και οι διαδικασίες. Πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε τέτοια δάνεια και πιστώσεις. Χρειαζόμαστε ταχύτατη δράση και δραστηριοποίηση. Πρέπει άμεσα να αντιδράσουμε σε αυτά τα θέματα. Πρέπει να δούμε την απάντηση στο ερώτημα επαρκούν όλα αυτά. Όχι, δεν επαρκούν. Πιστεύω ότι η σημερινή κατανομή και ταξινόμηση όσον αφορά τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη δεν επαρκεί για επαρκή διαφοροποίηση ώστε να διευκολύνεται η πρόσβασή τους σε κονδύλια. Κύριε Πίτροπε, θα πρέπει να προβληματιστούμε και να δούμε μήπως η πρακτική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα έπρεπε να αλλάξει. Μία πολιτική προκαταβολών που θα δίναμε θα ήταν κάτι καλύτερο. Θα βελτίωνε τις ε, προϋποθέσεις για την πρόσβαση στην αγορά, θα βελτίωνε την θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και αυτό θα ήταν θετικό, διότι θα μπορούσαν όλους τους άνεργους να τους απασχολήσουν οι μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις. Σε ευχαριστώ. Πρόεδρε, Επίτροπε, υποστηρίζω οποιαδήποτε μέτρα βελτιώνουν το περιβάλλον, το επιχειρηματικό για τις ΜΜΕ. Έχουμε πολλά προγράμματα για τις ΜΜΕ. Όμως λέμε πολλά λόγια, γράφουμε πολλά πράγματα για αυτές τις ΜΜΕ, δυστυχώς όμως τα αποτελέσματα είναι ισχνά. Πολύ συχνά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διευθύνονται από άτομα που έχουν ανεπαρκή κατάρτιση και εκπαίδευση. Χρειάζονται απλοί κανόνες και κανονισμοί λοιπόν για να είναι εύληπτοι για αυτούς. Τι πρέπει να γίνεται. Αν δεν αναγκάσουμε τις κυβερνήσεις μας να υιοθετήσουν υποχρεωτικά μη γραφειοκρατικούς κανονισμούς και κανόνες, τότε οι υπάλληλοι στις χώρες μας θα εξακολουθούν, θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν αυτές τις επιχειρήσεις ε, και να επιβάλλουν τις δικές τους απόψεις. Αν μπορούν να βρουν εκείνον τον οποίο θα μπορούν να ταλαιπωρούν θα χαίρονται ίσως κιόλα. Πιστεύω απόλυτα ότι η γραφειοκρατία είναι το κύριο πρόσκομα και εμπόδιο για αυτές τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια η κυρία Άγγελ. Αντζελίλη θα λάβει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν 24 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όλο ο παραγωγικό ιστό πάνω από 90% στην Ευρώπη και 98% στην ε, Ιταλία είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι συνήθως επιχειρήσεις με λιγότερο από 50 εργαζομένους, ακόμα και μικροεπιχειρήσεις με πολύ μικρότερο αριθμό. Δεν είμαι λοιπόν υπέρ αυτών που θέλουν να αυξήσουν τα, το κατόφλι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί έτσι θα επιδεινωνόταν ακόμα περισσότερο η πρόσβαση αυτών των επιχειρήσεων στην κοινωτική χρηματοδότηση. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε την πιο εύκολη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδίω στα διαδοτικά ταμεία, γιατί βρισκόμαστε σε μια φάση κρίσης όπου έχουν μεγάλη δυσκολία να πάρουν χρηματοδότηση. Είναι ιδιαίτερα επαχθεί και γραφειοκρατικές διαδικασίε και αποτρέπουν όλου αυτού του ε, δυνητικού ε, δικαιούχους. Η Γερμανία, η οποία είναι πάρα πολύ αποτελεσματική σε, στη χρήση των διαφορετικών ταμείων, έχει να αντιμετωπίσει τεράστια καθυστέρηση στην ε, χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Η κυρία Άντρες Μπαρέα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ του εκπροσώπους της Κομισιόν και του Συμβουλίου που συζητούν αυτό το θέμα μαζί μας και κατανοούν τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι απαραίτητο να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη. Έχουμε 25 εκατομμύρια μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κύριο δημιουργό θέσεων απασχόλησης. Χρειάζονται περισσότερες πιστώσεις και λιγότερη γραφειοκρατία. Το τέλος του Μαΐου θα έχουμε ένα συμβούλιο που θα ασχοληθεί Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα ασχοληθεί με την ε, απασχόληση και την ανάπτυξη. Τι θα κάνει λοιπόν για να έχει καλύτερη δυνατότητα πρόσβαση σε πίστοση η μικρομεσαία επιχειρήση. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνονται για την απασχόληση των νέων. Θα ήθελα το Συμβούλιο να μπορέσει ενώπιον μια τόσο σοβαρή κατάσταση να πάρει συγκεκριμένα μέτρα για όλα αυτά. Σα ευχαριστώ, Λεοπρόεδρο. Η κυρία Μαζέη Κουκόβιτς έχει το λόγο σε ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αξιότιμο κύριε Επίτροπε. Σήμερα ταχύτητα απαιτείται. Πρέπει γοργά να δράσουμε για τις επιχειρήσεις που δίνουν αγώνα για την επιβίωσή τους ε, και για την ανάπτυξή τους. Και βλέπουμε βραδύτερους ρυθμούς που υιοθετούνται από τα θεσμικά όργανα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όμως εξαρτώνται άμεσα από τη χρονική συνιστός, από την άμεση δράση που θα αναλάβουμε, δραστηριότητες άμεσες και απλούστευση. Πρέπει να τις ενθαρρύνουμε, να δώσουμε περισσότερες γνώσεις που θα διαχέονται, περισσότερες ευκαιρίες που θα δημιουργήσουμε, ακριβώς την εκπαίδευση, παιδεία, κατάρτιση. 60% των νέων μας δεν είχαν δυνατότητα μέχρι σήμερα να μετεκπαιδευτούν ή να επιμορφωθούν όσον αφορά τα θέματα επιχειρήσεων. 23 εκατομμύρια αυτές επιχειρήσεις δεν εκμεταλλεύονται όλους τους διάβλους ε, πληροφοριών και γνώσεων που είναι διαθέσιμοι. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι... πραγματικά η ραχοκοκαλιά. Η οικονομική κρίση είχε επιπτώσει ε, δραματικέ σε αυτή τη ραχοκοκαλιά που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση οι μικρομεσαίες επιχειρήσει, Μια και είναι η κύρια πηγή χρηματοδότηση, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση προ αυτέ τι επιχειρήσει και υπάρχουν τα ευρωπαϊκά μέσα για την υποστήριξή τους και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, πιστεύω πρώτον ότι είναι απόλυτα αναγκαίο αναγκαία επιταγή την επόμενη περίοδο να διατηρήσουμε αυτή την κατηγορία δράσεων για αυτές τις επιχειρήσεις. Δεύτερον, είναι αναγκαίο να έχουμε εθνικές και περιφερειακές αρχές που θα εμπλέκονται από την πρώτη φάση ήδη των μέτρων υποστήριξης και διαχείρισης νέων προγραμμάτων για το μέλλον, ώστε να υιοθετηθεί η πιο αποτελεσματική πολιτική μελλοντικά για την ενίσχυση των, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους. Η κυρία Φλασίκοβα Μενιώβα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, Επίτροπε, θα ήθελα να αναφέρω ότι σε σχέση με αυτή τη συζήτηση θα συμφωνήσουμε όλοι ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πραγματικά η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας απασχολούν τους περισσότερους εργαζόμενους και αυτό επειδή οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν συνήθως τις έδρες, έδρες τους σε ασιατικές χώρες ε, για λόγους ευνοϊκότερης φορολόγησης, για λόγους κόστους. Ελπίζω ότι θα μπορέσει να συζητηθεί αυτό το θέμα και στο μέλλον βέβαια. Η οικονομική κρίση έπληξε ιδιαίτερα βάναυσα ε, και επώδυνα τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, Αγωνίζονται να επιβιώσουν αυτή τη στιγμή. Είναι όμω ακόμα πιο επιτυχής ε, από ότι οι μεγάλε επιχειρήσει και προσαρμόζονται πιο εύκολα. Δυστυχώ είναι πολύ πιο δύσκολο οι μικρομεσαίε επιχειρήσει όμω να βρουν χρηματοδότηση από ότι για τι μεγάλε επιχειρήσει που δεν έχουν προβλήματα. Δεδομένη τη τεράστια σημασία των ΜΜΕ στην ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει να εξεύρουμε νέου τρόπου και μέσα να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια των διαθροτικών ταμείων. Πρέπει να άρουμε, να εξαλείψουμε τα γραφειοκρατικά εμπόδια και προσκόμματα και να διευκολύνουμε την πρόσβαση σε δάνεια και πιστώσει των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Λυπούμε, δεν μπορώ να δω πώ πάει το ρολόι, αλλά μια και μου λέτε ότι θα πρέπει να σταματήσω, σταματώ πρόεδρε. Ευχαριστώ. Εσύ συνέχεια, εσεί κυρία έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συναδελφοί. Τα μέσα ενημέρωσης φαίνεται να ανακαλύπτουν τώρα την ανάγκη να έχουν μια μακροχρόνια στρατηγική ανάπτυξη, ενώ αυτό ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό ο πυρήνα τη οικονομική μα στρατηγική. Είναι απαραίτητο να υπάρξει και καλύτερη χρησιμοποίηση των δημοσίων πόρων και κατεύθυνσή τους προς επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις απασχολήσεως, δηλαδή κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα 23 εκατομμύρια μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη είναι ζωτικά εργαλεία για την ανάπτυξη και τη χωροταξική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Αλλά έχουν μεγάλες δυσκολίες για να βρουν χρηματοδότηση και η τωρινή κρίση κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Το Φεβρουάριο είχαμε ήδη συζητήσει το θέμα της χρήσης των διαφορετικών πόρων για να αντιμετωπίσουμε την αργία των νέων και να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η έκθεση του Ελεκτρικού Συνεδρίου το Μάρτιο μας κατέδειξε αυτό το οποίο πιστεύαμε από πάρα πολύ καιρό. Ότι είναι πολύ πολύπλοκα τα εργαλεία ε, χρηματοοικονομικής μηχανικής για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους. Πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε και να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση που αφορά ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι γνωστές οι δυσκολίες τους. Είναι ο καιρός να κατανοήσουμε καλύτερα την πολυπικιλία των αναγκών τους μέσα στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Σε ευχαριστώ όλους τους ομιλητές και θα δώσω τώρα το λόγο στον Επίτροπο Χάν. Σε ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Στον χρόνο που έχω δυόμιση λεπτά δεν είναι δυστυχώ δυνατόν να επιστρέψω σε όλα τα θέματα που εκκρεμούν και τις παρεμβάσεις σας. Θα δοθούν γραπτώσει οι απαντήσεις μου. Όμως οι κυριότερες κατηγορίες ε, των ερωτήσεών σας για την τρέχουσα περίοδο πρώτα. Ναι, εδώ υπάρχουν ε, αναδιαρθρώσεις και δράσεις, όμως τα κράτη-μέλη είναι εκείνα τα οποία πρέπει να υποβάλουν τις αντίστοιχες προτάσεις. Να είσαστε βέβαιοι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη όλες αυτές τις προτάσεις, όχι μόνο με θετικό πνεύμα, αλλά και με ιδιαίτερα θετική αντιμετώπιση και δράση, ώστε να καταπολεμηθεί η ανεργία, ιδιαίτερα η ανεργία των νέων, με αυτά τα μέτρα που θα λάβουμε. Παρακαλώ να δώσετε την υποστήριξή σας στα κράτη-μέλη σας σε αυτές τις δράσεις ή στις εκλογικές σας περιφέρειες να μας υποστηρίξετε σε αυτές τις πρωτοβουλίες μας. Συχνά αναφέρθηκε για τη μελλοντική υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τι πρέπει να γίνει. Για τη μελλοντική περίοδο προγραμματισμού, σχεδιασμού έχουμε ένα ελάχιστο πλαίσιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προβλέπετε. Στην εισαγωγή μου είπα 80% ουσιαστικά για τις ε, πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες, 50% για τις λιγότερο ανεπτυγμένες. Όμως παρακολουθώ και τη συζήτηση στην Ευρωβουλή, όπου αυτά τα όρια έχουν ε, υποστεί επικρίσεις και παρακαλώ αν πραγματικά πιστεύετε ότι εμείς στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουμε στην καινοτομία τους και την ε, δυνατότητα καινοτόμα να δρουν, πρέπει να συνεισφέρετε και εσείς από πλευρά σας. Αυτές οι ελάχιστες ε, προσπάθειες ε, με κονδύλια να διασφαλιστούν. Τελικά είναι αναγκαίο να βρούμε κομμένες και ραμμένες ειδικά για τις ανάγκες τους λύσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε σχέση με τα διαθέσιμα κονδύλια και τα διαθέσιμα μέσα ώστε να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Και ιδιαίτερα για εκείνους που ασκούν κάποιες επικρίσεις και λένε ότι στο ένα ή άλλο σημείο η υλοποίηση όσον αφορά και τα κονδύλια και την μεγάλη γραφειοκρατική επιβάρηση και χρονική υπερβολική διάρκεια μέχρι ότου να υποφεληθούν οι τελικοί αποδέκτες θα πρέπει και εμείς να δράσουμε να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση να μην είναι πλέον έτσι τα πράγματα στο μέλλον αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις ότι αν εκείνο το πλαίσιο του μελλοντικού πλαισίου ε, που αφορά την ανάπτυξη την αηφορία στην ανάπτυξη αν εστιαστούμε σε αυτό με 500 ε, δισεκατομμύρια που θα προβλεφθούν τότε θα πρέπει πριν από το καλοκαίρι να μπορέσουμε να αποσαφηνίσουμε και να πούμε ότι αυτά τα κονδύλια στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο θα είναι διαθέσιμα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα δίναμε ένα σαφέστατο μήνυμα προς τους πολίτες της Ευρώπης και όλοι θα γνώριζαν ότι υπάρχει προγραμματισμός και ασφάλεια προγραμματισμού προς ποια κατεύθυνση θα υπάρξουν επενδύσεις και υποστήριξη. Θα μπορούσα να πω ότι με αυτόν τον τρόπο θα αναπτυχθεί μια όθηση, ένα νέο κύμα όθησης και υποστήριξης που θα είναι υποφελές για την ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Thank you. And finally, Mr. for Council κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι βουλευτέ, η συζήτηση σήμερα. Η σημερινή συζήτηση έχει εστιάσει στο θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την πρόσβασή του σε χρηματοδότηση καθώ και το θέμα του ορισμού του λόγω της ε, οικονομική κρίση είναι ιδιαίτερα επίκαιρο αυτό το θέμα. Εγώ θέλω να υποστηρίξω αυτά που ελέγχθησαν υπέρ τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι ουσιαστική και ζωτική για να μπορέσουν να επιβιώσουν μέσα σε αυτό το κλίμα μικρομεσαίε επιχειρήσει. Είναι γνωστό ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην καινοτομία και στην δημιουργία απασχόληση. Μα ενδιαφέρει ιδιαίτερα από τη Δανική Προεδρία να εξασφαλίσουμε τη δημιουργία μια αγορά κεφαλαίου κινδύνου για τα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη δημιουργία ενός πιο έφορου κλίματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να υπάρξει δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξη. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλου αυτού οι οποίοι έλαβαν το λόγο, ιδιαίτερα τον κύριο Μπένσεν και την κυρία Κρέελ. Έχω τονίσει, θέλω να τονίσω ότι έχετε τονίσει ιδιαίτερα την δημιουργία, την ανάγκη δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση και τον ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ε, αποδοτική χρήση της ενέργειας. Αυτά είναι θέματα τα οποία βρίσκονται και στην καρδιά της προσπάθειας της ε, Δανικής Προεδρίας, η οποία δίνει συνέχεια στην, ε, στο Small Business Act, στην νομοθεσία αυτή του 2008 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, Αναφέρθηκε η ανάγκη να υπάρξει μια ενσωμάτωση τη προβληματική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλε τι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρξει μια ε, απάλυνση και απλοποίηση των διαδικασιών που τι αφορούν. επίση να υπάρξει και μια πραγματική πρόοδο στο ψηφιακό θεματολόγιο προ την κατεύθυνση και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τρίτο, και αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο θέλω να δώσω μια απάντηση στον κύριο Ρίμπιξ, στον κύριο Κάλφιν και στον κύριο Φανίστ Λερόι, ένα σημαντικό στοιχείο Τη διαπραγμάτευση του δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 θα πρέπει να είναι η εστίαση σε περισσότερη ανάπτυξη αλλά και αυτό αφορά και τη χρησιμοποίηση των διαφορετικών πόρων που θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτή τη στρατηγική. Και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο της Δανικής Προεδρίας και των προοπτικών της που δίνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το πλαίσιο. Θέλω λοιπόν για όλα αυτά να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, συζήτηση αυτή και θέλω να σας τονίσω ότι όλοι μαζί Κομισιόν, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο θα μπορέσουν να προωθήσουν τα θέματα αυτά ώστε να μπορέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης και πάλι να ανθίσουν και να δώσουν θέσεις απασχόλησης σε όλους αυτούς τους νέους οι οποίοι περιμένουν συγκεκριμένα και αυτά αποτελέσματα από μας. Ευχαριστώ. Thank you, Thank you, Council. Thank you, colleagues. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε συνάδελφοι. Η συζήτηση περαιώθηκε. Περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη τώρα. Δήλωση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είπα της εκπρόσωπους για την κατάσταση στην εξωτερική πολιτική, για την κατάσταση στην Ουκρανία όσον αφορά την Γιούλια Τιμοσέγκο. Είπατε